δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ο, η πρώτη ομιλήτρια εξ ονόματος του Συμβουλίου είναι η Υπουργό Τζάντα Κάλνινα Λουκασέβιτσα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδεται να ασχοληθώ με το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ε, υποχρεούμεθα να διασφαλίσουμε για τους πολίτες έναν χώρο πραγματικής ελευθερίας και δημοκρατίας και ασφάλειας, καταπολεμώντας το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα μας τα μέσα και εργαλεία για αυτό το σκοπό και να ενώσουμε τις προσπάθειες για μια συνεκτική και σφαιρική προσέγγιση απέναντι στο έγκλημα. Η Europol υπολόγισε στην έκθεσή της για το, του 2013 ότι 3.000 600 ομάδες οργανωμένου εγκλήματος δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκληματικές οργανώσεις ε, που επιδεικνύουν μεγάλη ευελιξία και διαφοροποιούν τις δραστηριότητες τους. Ε, συνεχώς ε, αυξάνονται καλύπτοντας όλο και ευρύτερο φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων, ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση τεχνολογικών ε, εξελίξεων κλπ. Ε, δημιουργούνται τεράστια κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες ε, που περνούν στην πραγματική οικονομία. Οι εγκληματικές ομάδες όλο και περισσότερο μπορούν να επηρεάζουν τη λειτουργία των νόμιμων αγορών και ακόμα και τα θεσμοί, οι θεσμοί και οι πολιτικές διαδικασίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, επηρεάζονται από τις πρακτικές της διαφθοράς. Το Συμβούλιο συνεχώς ε, συμμετέχει σε σειρά δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και τα αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητα. Αξιότιμα μέλη, ένα κέριο μέτρο είναι ο κύκλος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε το 2010 και διασφαλίζει επιχειρησιακή απόκριση στο σοβαρό οργανωμένο διεθνές έγκλημα μέσα από βέλτιστο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαίων, ε, εθνικές ε, ε, μονάδες επιβολής δικαίου και άλλους εμπλεκομένους. Το Συμβούλιο συμφώνησε γι' αυτό σε μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων που στοχεύουν μεταξύ άλλων ε, στην παραχάραξη, στο κυβερνοέγκλημα που ε, συμφωνήθηκε ότι είναι προτεραιότητες ε, στο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορία αγριών ζώων, εμπορία πολιτιστικών αγαθών, Εντοπίστηκε επίσης από το Συμβούλιο ως τομείς που χρήζουν προσοχής. Τέτοια εγκλήματα θα παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από τη Europol που αναμένεται να υποβάλει στο Συμβούλιο μία ενδιάμεση ε, αξιολόγηση για το οργανωμένο έγκλημα ε, το Μάρτιο του 2015. Το Συμβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην έκθεση καταπολέμησης διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Φεβρουαρίου του 2014. Πρόκειται για πολύτιμο εργαλείο που θα ενοποιήσει τις προσπάθειές μας και θα προωθήσει πρότυπα υψηλά η καταπολέμηση διαφθοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στη βάση μιας σφαιρικής προσέγγισης. Πιστεύουμε ότι θα δοθούν έτσι περισσότερα κίνητρα στα κράτη-μέλη για να ε, επικυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα μέσα καταπολέμησης διαφθοράς που υπάρχουν. Ο ρόλος της ανάκτησης των κεφαλαίων ή κερδών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της μάχης κατά του διασυνοριακού οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος. Οι εγκληματικές ομάδες μπορούν να συσσωρεύουν τεράστια κέρδη από διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες στις αγορές και γενικά συμφωνούν όλοι ότι η ανάσχεση των ε, κινήσεων των κλιματικών ομάδων είναι ένα σημαντικός τρόπος ε, για να μειωθούν τα έσοδα από τις εγκληματικέ δραστηριότητε. Η νέα οδηγία για το πάγωμα και τη δίμευση των προϊόντων από παράνομε δραστηριότητε που εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2014 ε, δίνει ευρύτερες δυνατότητες για τη δίμευση των προϊόντων του εγκλήματος σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη γιατί ε, ο ύποπτος ε, ρημοδική ε, έχει διαφύγει. Επίσης προβλέπεται ένα ενισχυμένο σύστημα ευρύτερης δίμευσης η δίμευση και από τρίτον. Αυτό το μέσο είναι ένα πολύ καθαρό βήμα μπροστά γιατί διασφαλίζει ότι οι εγκληματίες δεν θα έχουν πια πρόσβαση στα κέρδη που ε, προέρχονται από κάποιες ε, κατηγορίες εγκληματικών δραστηριοτήτων και αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της απο, απόκρισης σε σοβαρές μορφές εγκλήματος. Κατά τις διαπραγματεύσεις ε, μέχρι την έγκριση αυτού του μέσου, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα σε αυτό το τομέα. Και γι' αυτό το σκοπό ενέκριναν μαζί με την οδηγία και δύο δηλώσεις που καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής περαιτέρω προτάσεων επί του θέματος αυτού. Το Συμβούλιο προσβλέπει στην, στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το θέμα. Τέλος. Ε, επιτρέψτε μου να σχολιάσω εν συντομία την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Πρόκειται για υψηλή προτεραιότητα, υψηλής θέμα για το Συμβούλιο. Θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ζητάει αναθεώρηση και ενημέρωση της εσωτερικής στρατηγικής ασφάλειας μέχρι το μέσον του 2015. Πέρσι το Δεκέμβριο το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα τα οποία ε, παρουσιάζουν τις σκέψεις του Συμβουλίου ε, πάνω στο γενικότερο θέμα και κάποιες βασικές αρχές σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της Ένωσης για την ασφάλεια. Μια βασική αρχή είναι ότι η ανανεωμένη αυτή στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να εντοπίζει τις βασικές απειλές και προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα σε όλες τις μορφές του συνιστά μια από αυτές τις απειλές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Υπουργέ που μιλήσατε εξ ονόματος του Συμβουλίου. Και τώρα ε, καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και πάλι και του δίνω το λόγο ε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, διότι μου δίδεται την ευκαιρία να παρουσιάσω την πολιτική και τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα για την ανανέωση της ε, εσωτερικής στρατηγικής ασφαλείας, ε, το οποίο υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου καλώς τονίζει τις προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να προωθήσουμε ε, και στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουμε ε, τη δουλειά μας τα επόμενα χρόνια. Καταπολεμώντας ε, αυτή τη μάστιγα με όλες τις, δυνάμει, δυνάμεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει μια πιο ασφαλή ήπειρο αν θέλετε, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. η καταπολέμηση της παρίσφρησης του οργανωμένου εγκλήματος στην πραγματική οικονομία θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην ανάπτυξη. Και αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ για τη διαφθορά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν για τη ε, διαφθορά. Στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου ε, το 2013 φάνηκε ότι άνω του μισού των Ευρωπαίων πολιτών ε, θεωρούν ότι η διαφθορά στην εκάστοτε χώρα, τη δική τους, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τέσσερις στις δέκα ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί τροχοπέδι για το επιχειρήν στην εσωτερική αγορά. Η πρόληψη λοιπόν της διαφθοράς και η προώθηση της ακαιρεότητας της εντιμότητας είναι κάτι που έχει ανέβει στην κατάταξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την τελευταία δέκα ετία. Ε, σύμφωνα με τις εκθέσεις, ε, η διαφθορά σε μία χώρα και η ε, επέκτασή της σε άλλες χώρες είναι κάτι που τελικά πλήττει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Σίγουρα είναι σημαντικό να έχουμε σωστή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, σχετικών διεθνών θεσμικών οργάνων. Η επόμενη έκθεση ε, θα, για το θέμα αυτό θα συνταχθεί επισήμως το 2016 και στη δεύτερη έκθεση υπάρχει έτοιμα να συμπεριληφθεί ο στόχος η ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα το εξετάσουμε αυτό ε, έχοντας ε, διαβουλευθεί με τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ε, θα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει μέτρα για να αυξήσει τη δική της διαφάνεια και η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την πρόληψη της διαφθοράς. Έρχομαι τώρα στο οργανωμένο έγκλημα. Για να πω ότι είναι σαφέστατο το πόσο σοβαρό είναι. Αυτό τεκμεριώνεται στην ετήσια έκθεση της Europol. 3.000 ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ε, σε πολλά είδη ε, αδικημάτων. Περιλαμβάνεται εκεί το οικονομικό έγκλημα, το ξεπλήμα χρήματος, το κύβερνο έγκλημα ή και το περιβαλλοντικό έγκλημα. Οι επενδύσεις του οργανωμένου εγκλήματος είναι όλο και πιο διεθνείς και έτσι το οργανωμένο έγκλημα παρισφρεί στην πραγματική οικονομία ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί στο έπακρο. Και αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για την απόφαση πλαίσιο του 2008 για την καταπολέμηση του εργονομένου εγκλήματος. Μία απόφαση πλαίσιο για την οποία θα συντάξει έκθεση εφαρμογής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος, ή αυτή τη χρονιά. Η οδηγία που υιοθετήθηκε πέρσι για τη δίμευση και την κατάσχεση, το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικού είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η πρόσφατη συμφωνία για την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων προσόδων είναι πολύ σημαντική. Περιλαμβάνονται δράσεις για να εντοπιστούν πιο εύκολα οι δικαιούχοι, αυτοί που ωφελούνται τελικά από την αλυσίδα αυτή της παραβατικής δραστηριότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέσω της Europol ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών αλλά και μεταξύ των χωρών μελών και τρίτων χωρών. Οι προτεραιότητες της ε, Europol περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την λαθρομετρία μετανάστευση, την, το, τη διακήρυξη ανθρωπίνων όντων, τα παραποιημένα, ε, τα, πλαστο, ε, τα παραποιημένα προϊόντα, της τις ε, παραβάσεις για, σε σχέση με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πυροβόλων όπλων, το λαθρεμπόριο όπλων, μεταξύ άλλων. Χρηματοδότηση ε, γίνεται μέσω του, του Ταμείου για την Εσωτερική Ασφάλεια. Ένα δις περίπου για την περίοδο 2014 με 2020. Έτσι χρηματοδοτούνται οι δράσεις μας. Και ε, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο λαθρεμπόριο όπλων κατόπιν και των τραγικών ε, γεγονότων ε, της περασμένης εβδομάδας. Η Ευρωπόλ, η Europol το έχει εντοπίσει αυτό το, αυτή την παράνομη δραστηριότητα ως μια αναδυόμενη απειλή που θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόμενο να προτείνει να προτείνει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για ορισμένες κατηγορίες πυροβόλων όπλων, να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τα, την παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων. Σε κάθε περίπτωση η πρόληψη είναι η πιο ισχυρή συνιστόσα της μάχης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπλέκουμε ενεργά τις τρίτες χώρες και ε, τα διεθνή θεσμικά όργανα. Έχουμε μια πολύ γεμάτη ατζέντα στη συνεργασία μας με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες για το κυβερνοέγκλημα και την παιδική κακοποίηση. Με τους εταίρους μας προς Ανατολάς δίνουμε έμφαση στη διαφθορά. Η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος ε, είναι βασική προτεραιότητα σε σχέση με την στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια. γιατί <coughs> είναι κάτι που πλήττει και επηρεάζει την οικονομία, τους πολίτες, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν για παράδειγμα υποκλέπτονται προσωπικά δεδομένα πελατών ή εργαζομένων πολιτών και όταν ε, χάνονται περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε ε, δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Κυβερνοεγκλήματος μέσα στην Europol και θα πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να ε, υλοποιήσουν σχετικές δράσεις μέχρι το Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς. Καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι το σχέδιο οδηγίας για την ασφάλεια των πληροφοριών και ούτω καθεξής θα περιλάβει διατάξεις για την αναφορά τέτοιων συμβάντων κυβερνοεγκλήματος στις ε, διοκτικές αρχές. Αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, οι ε, ε, για να ε, η έρευνα και η ανάκριση και όλη αυτή η διερευνητική δραστηριότητα σε περίπτωση κυβερνοεγκλήματος είναι κάτι που πρέπει και μπορεί να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, είναι έτοιμη να το κάνει έτσι ώστε η φυστάμενη νομοθεσία για τις κυβερνοεπιθέσεις και για τις απάτες της πληρωμές και για την παιδική κακοποίηση, τη διαδικτυακή, όλα αυτά, ε, όλες οι διατάξεις για την καταπολέμηση όλων αυτών ενσωματώνονται γρήγορα και εφαρμόζονται ε, στο έπακρο. Η συνεργασία μας ασχολ... έχει να κάνει επίσης και με τις προκλήσεις ε, που ε, περιλαμβάνει η δυνατότητα και η υποχρέωσή μας να αφαιρούμε παράνομο περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Ε, και η συνεργασία έχει να κάνει και με την καταπολέμηση των τρομοκρατικών ενεργειών μέσω διαδικτύου. Η συνεργασία ε, με εσά είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε ομαλά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Σα ευχαριστώ θερμά. Η πρόεδρο, ευχαριστώ. Θα κάνουμε τον ε, γύρο των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Χολμάιερ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, στην πάλη κατά του οργανωμένου εγκλήματος μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική πολιτική της. Γιατί το έγκλημα μπορεί να δικτυώνεται, μπορεί να υιοθετεί βάναυσους και ομούς τρόπους ε, μεθοδεύσεων και πάντοτε βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τα μέτρα τα δικά μας. Γι' αυτό πρέπει να ζοριστούμε πολύ, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα στην πολυσχηδή του δράση. Έχω υπόψη μου εδώ κυρίως το διαδίκτυο, όπου υπάρχουν πάρα πολλές μορφές εγκλήματος που μαζικά συνεχίζονται μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, ε, πορνογραφία παιδική. Ε, εκεί, μέσα από το διαδίκτυο, είδαμε μια τεράστια αύξηση. Ο αριθμός των παιδιών που πλήττονται έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη χώρα τη δική μου. Και βέβαια ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να συζητήσουμε, παρόλο που δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, πρέπει να δούμε τις ε, τελευταίες έρευνες σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Ε, πολλές φορές η αδράνεια δρά ως καταλήτης ε, και οι εγκληματικές δραστηριότητες ε, αυξάνονται και πληθύνονται. Νομίζω ότι τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, αλλά η στρατηγική αυτή δεν εξαντλείται εδώ. Πρέπει να επανέλθουμε πολλές φορές σε αυτήν και να τη συζητήσουμε εντελεχώς. Δέχεστε μια μπλε κάρτα, κυρία Χολμάιερ, από τον κύριο Σάνι. 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. nagyon Σας ευχαριστώ πολύ. Να βοηθήσω λίγο την κυρία Χολμάιερ, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να αφαιρθεί σε όλα τα φαινόμενα. Αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα και η διαφθορά αποτελεί βέβαια μέρος της εγκληματικότητα. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας, κυρία Χολμάιερ, όσον αφορά την οργανωμένη μορφή της διαφθοράς και όταν υπεύθυνο για το φαινόμενο αυτό είναι το ίδιο το κράτος μέλος, η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους. Αγαπητέ συνάδελφε, η διαφθορά είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι η προσπάθεια άσκηση πίεσης στην πολιτική. Μέσα από τη διαφθορά ανοίγει δρόμους. Και όταν το καταφέρουν και εδρεωθούν, εμείς πρέπει να τους απομακρύνουμε με όλες τις δυνατότητες που μας δίνουν τα διαθέσιμα μέσα και ε, ε, εργαλεία. Προφανώς είναι πάρα πολύ ασυμμορφές της διαφθοράς. Η κυρία Κίνιτσι, εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, να ευχαριστήσω επίσης την εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην εργασία της Ιταλικής Προεδρίας στο τελευταίο εξάμεινο, όπου ουσιαστικά δεν κατάφερε να προχωρήσει πάρα πολύ και εξαιτία της ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο νομίζω ότι τα νομοθετήματα τα οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή όπως η οδηγία PIF για το οικονομικό έγκλημα αλλά καθώς επίσης και άλλες οδηγίες είναι πάρα πολύ σημαντικές προκειμένου να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα καθώς επίσης και τη δραστηριότητα των μαφιόζικων οργανώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να λάβουμε υπόψη μας επίσης και τα συμπεράσματα της συνεργασίας για την ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά τον τομέα των τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε όμως να καταλήξουμε σε μία να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε την απόφαση πλαίσιο του 2008 για το οργανωμένο έγκλημα. Έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια από τότε και νομίζω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τα μέτρα εκείνα που έχουν να κάνουν με την κατάσχεση και την ανάκτηση των προϊόντων του εγκλήματος. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πιο φιλόδοξη πρόταση όσον αφορά τη δέσμευση, κατάσχεση και ανάκτηση των προϊόντων του εγκλήματος, καθώς επίσης και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την καταδίκη των δραστών των εγκληματικών πράξεων. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πατάξουμε την εγκληματικότητα σε όλες τις μορφές της. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό τμήμα της δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Φοϊβόσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο περίεργο να μιλάμε για διαφθορά και παράλληλα για εγκληματικές ε, δραστηριότητες εν γέννη. Θα έπρεπε κανονικά τη διαφθορά να την αντιμετωπίσουμε ως ξεχωριστό φαινόμενο. Έχει να κάνει κυρίως με αυτούς οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την εξουσία. Αν τα θεσμικά όργανα λειτουργούν σωστά, τότε δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για την εμφάνιση της διαφθοράς. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε για διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των μεμονωμένων κρατών μελών. Και πολύ συχνά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο διαφάνειας. Μέσω της διαφάνειας μπορούμε να προλάβουμε την εμφάνιση της διαφθοράς. Στην Πολωνία πολλές φορές δεν καταφέρνουμε τελικά να δούμε ποιος και κατά ποιο τρόπο χρησιμοποίησε κάποια κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υλοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να καταλήξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όταν δεν έχουμε τα δεδομένα αυτά. Κυρία ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, πριν από ένα χρόνο εγκρίναμε μια ειδική έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα που περιείχε κάποιες συστάσεις. Για παράδειγμα, ενίσχυση το, του Frontex και ε, δικαιώματα θυμάτων, προγράμματα προστασίας κλπ. Ε, θέλω να ρωτήσω την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο προχωρήσατε σε σχέση με την εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας επέτρεψε καλύτερη συνεργασία μεταξύ αστυνομιών και δημοσίων αρχών, αλλά χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία μας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων, για παράδειγμα. Η Eurojust, η Europol ε, μπορούν να ε, δρούν καλύτερα, ε, με καλύτερη οργάνωση. Πρέπει επίσης να προβλέψουμε νομική προστασία για τους ανηλίκους. Ε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση, την προστασία των πολιτών μας πάνω στη βάση της, των αναγκών, της αναλογικότητας και τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από αυτό σήμερα που ζούμε στη σκιά του σοκ από τις επιθέσεις στο Παρίσι. Κουνσάλεφ Πένιασε, Τάνια, εξ ονόματος του Αριστεράς. Μιλούμε για διαφθορά και δεν μιλούμε για πολιτική διαφθορά. Αναρωτιέμαι. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βάζουμε τη διαφθορά ε, στο ίδιο θέμα με το οργανωμένο έγκλημα. Επειδή δηλαδή δεν θέλουμε ουσιαστικά να μιλήσουμε για την πολιτική διαφθορά. 40 δις ευρώ ε, στοιχίζει αυτό το σύστημα διακυβέρνησης το διεφθαρμένο που έχουν δημιουργήσει ε, τα μεγάλα κόμματα ε, της καθεστικίας τάξης και δεν μιλούμε μόνο για ξέπλυμα χρήματος αλλά και για τα τεράστιες, για τις μίζες και όλα αυτά, όλες αυτές τις απάτες αλλά μιλούμε και για τα νομικά συστήματα που επιτρέπουν να υπάρχει φοροδιαφυγή από πλευράς επιχειρήσεων. Θα πρέπει να γίνει ε, ε, διερευνητική επιτροπή εναντίον των ηθινόντων και ε, λείπουν 14 υπογραφές από τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας για να μαζέψουμε τις υπογραφές και ε, να γίνει η ερευνητική ε, διαδικασία. Ο κύριος Γιαβόρ, εξ ονόματος των Πρασίνων, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στι παρεμβάσει μα και ακριβώ επειδή οι παρεμβάσει είναι αρκετά αποτελεσματικέ εξ ονόματο Επιτροπή και του Συμβουλίου, υποβάλαμε εμεί ένα προφορικό ερώτημα. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική στρατηγική κατά τη διαφθορά προκειμένου να καταφέρουμε να συσπυρώσουμε, να συντονίσουμε τις διάφορες οδηγίες και τους διάφορους κανονισμούς που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε όμως και μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να καταφέρουμε να καταβάλουμε πιο σημαντικές προσπάθειες πολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Αν δεν λάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, τότε θα ζημιώσουμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα από, τη, από το Ταμείο Συνοχής τελικά θα καταλήξουν στι τσέπε των ολιγαρχών και στις τσέπες διαφόρων επενδυτών. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει και λιγότερο ελκυστική και όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Η κυρία Φεράρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής και θα έλεγα κάπως περήφανη που το ζήτημα της καταπολέμησης, διαφθοράς και της μαφίας έχει επιστρέψει και απασχολεί πλέον της, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στην πρωτοβουλία του κινήματος των πέντε αστέρων και χάρη στην συμβολή διαφόρων συναδέλφων από διάφορες χώρες. Θα ήμουν όμως ακόμα πιο ικανοποιημένοι αν οι Ιταλοί συνάδελφοι από το PD, το Δημοκρατικό Κόμμα δηλαδή, είχαν καταφέρει να παραμερίσουν τις κομματικές τους διαφορές και μας είχαν τελικά υποστηρίξει, πράγμα το οποίο δεν κάναν και αυτό αποτελεί ξεκάθαρη ντροπή και νομίζω ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, οι συναδελφοί μου δηλαδή από το PD, να θεωρούν αυτού πρωταθλητέ τη καταπολέμηση τη μαφία. Το οργανωμένο έγκλημα, η μαφία και η διαφθορά αποτελούν καρκίνωμα που καταστρέφει τελικά την οικονομία, την πολιτική, καθώ επίση και τι κοινωνικέ δομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο αυτό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ιδέα αυτή τη προφορική ερώτηση που μυστηριωδώ έγινε τελικά δήλωση του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση που σταμάτησε τον Οκτώβριο το 2013 όταν εγκρίναμε την έκθεση της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να συνεχίσει το έργο της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη θα πρέπει να εγκρίνει νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να πάρει μια απόφαση όσον αφορά το ζήτημα της σύμπραξης σε μια οργάνωση τύπου μαφίας και να θεωρηθεί αυτό έγκλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να προωθήσει περισσότερο τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος καθώς επίσης και να εισάγει μέτρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την καθυστερημένη κατάσχεση και τις καθυστερημένες συλλήψεις που αυτό απαιτείται για τη συλλογή των αποδεκτικών στοιχείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης το Συμβούλιο να αναλάβει επικοδομητική δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θέλω να πω ότι η Ιταλική Προεδρία δεν έκανε απολύτω τίποτα και δεν έδωσε καμία συνέχεια στα πορίσματα της Επιτροπής Κρίμα. Και βλέπουμε ότι επίση το PD του Ρέντσι δεν προωθεί καθόλου το προφορικό αυτό ερώτημα, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι για τον κύριο Ρέντσι και για το PD η καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο δεν αποτελεί προτεραιότητα. Κύριο Φουντούλη, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Πρόεδρε, αδελφοί, για το θέμα τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη διαφθορά, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν νόμοι στα κράτη-μέλη και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο το θέμα είναι εάν εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παρεμβάσεις. θα σας θυμίσω το σκάνδαλο της siemens στην ελλάδα εκατομμύρια ευρώ πήγαν στις τσέπες πολιτικών για μίζες προκειμένου η εταιρεία να έχει πρόσβαση στις κρατικές προμήθειες και επιλεκτική αντιμετώπιση εναντί των ανταγωνιστών της τον άνθρωπο της siemens στην ελλάδα τον κύριο χριστοφοράκο ο οποίος κανόνιζε τον χρηματισμό πολιτικών προσώπων όπως προέκυψε από τη διερεύνηση του σκανδάλου ενώ εναντίον του εκδόθηκαν συνολικά τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης η γερμανία ουδέποτε τον παρέδωσε στις ελληνικές αρχές για να δικαστεί προστατεύοντας φυσικά την γερμανικών συμφερόντων siemens. με τον τρόπο αυτό προστάτευε και κάποιους πολιτικούς από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στην ελλάδα όπως ο ίδιος ομολόγησε στην εισαγγελέα του μονάχου το 2009 ότι του έδινε χορηγίε για την καλλιέργεια του πολιτικού τοπίου. κύριοι συνάδελφοι ψηφίζουμε νόμους και ευρωπαϊκές οδηγίες τους εφαρμόζουν όμως όπως οφείλουν όλα τα κράτη μέλη. σας ευχαριστώ. Euh, Η κυρία Μακοβέ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται από το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά, την τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρήματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατία χρηματοδοτείται πάντα μέσω του οργανωμένου εγκλήματος και των οργανώσεών του. Εκατομμύρια ευρώ χάνονται ετησίως λόγω των εγκλημάτων αυτών και επειδή το βρώμικο χρήμα δεν δημεύεται και δημιουργεί νέα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό είναι σημαντική η καταπολέμηση αυτής της μορφής εγκληματικότητας. Να θυμίσω την οδηγία για την δίμευση και την εξωτερική δίμευση και τη δίμευση από τρίτους και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας σε κάθε κράτος μέλος είναι σημαντική και πρέπει να εφαρμόζεται επακριβώς για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, ε, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει να, με, τη μελέτη που υπεσχέθη σχετικά με τα κέρδη από τις εγκληματικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι η δίμευση στην αστική διαδικασία που ακολουθείται από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ χρήσιμη. Αν δεν προβούμε στη δίμευση των προϊόντων εγκλήματων, κάθε έρευνα στερείται νοήματος. Διακοπή. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Χόλτσερ. Το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά βλάπτουν το μέλλον και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή κάθε χώρας. Βέβαια, πρωτίστως είναι καθήκον των κρατών μελών να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι ένας κοινό χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης δικαι... και ε, ασφάλειας και έτσι ε, όλοι ενεχόμεθα στη διαδικασία καταπολέμησης. Ε, άλλωστε το, το οργανωμένο έγκλημα είναι διασυνοριακό. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει ε, εντονότατα να φροντίσουμε ούτως ώστε ε, να... Ε, ε, αναστείλουμε και καταστήλουμε τις δραστηριότητες αυτές. Πολλά κράτη-μέλη κατά το παρελθόν στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν οικονομικά ε, πλεονεκτήματα ε, φέρθηκαν με χαλαρότητα απέναντι στην φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Δημιουργήθηκαν φορολογική παράδειση που βέβαια είναι φυτόριο για εγκληματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασισμένοι εναντίον όλων αυτών. Ε, είναι πολύ σημαντική η νομοθεσία που θα ψηφίσουμε ε, στον τομέα αυτών. Θα πρέπει η μάχη να γίνεται με αποφασιστικότητα και πάντοτε θα πρέπει να φροντίζουμε παράλληλα ε, να διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί μόνο έτσι μπορεί να προσβλέπει κάθε κοινωνία στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Τόμασιτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι εγκληματικέ οργανώσει αποτελούν μια όλο και μεγαλύτερη απειλή για τα κράτη-μέλη. Διαταράσσουν την τάξη, διαταράσσουν την οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια και πολλέ φορέ χρηματοδοτούν του ίδιου του τρομοκράτε. Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι για μας να συνεργαστούμε για να πατάξουμε το οργανωμένο έγκλημα. Πραγματικά σοκαρίστηκα το γεγονό ότι ακούστηκε σήμερα στα μέσα μαζική ενημέρωση ότι οι σφαίρε που χρησιμοποίησαν οι δράστε των εγκλημάτων στο Παρίσι ερχόντουσαν από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε την απαραίτητη συνεργασία στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό θα γίνει αν επιτόπου αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση και αν καταφέρουμε τελικά να μειώσουμε τη γραφειοκρατία μα, αν καταφέρουμε ουσιαστικά να απλουστεύσουμε το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε του πολίτε μα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς έχει μείνει ουσιαστικά γράμμα νεκρό, διότι δεν υπήρξε πολιτική βούληση για την αποτελεσματική υλοποίησή του. Εκτός όμως από την καταπολέμηση της διαφθοράς στο μέλλον, πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες της διαφθοράς στο παρελθόν. Ένα μέρος της υπερχρέωσης πολλών κρατών μελών της Ένωσης οφείλεται στο ότι διεφθαρμένοι πολιτική ανέθεταν ιδίως σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ανώφελα στην ουσία δημόσια έργα και προμήθειες σε διονγκωμένε τιμές επιβαρύνοντας έτσι τους εθνικούς προϋπολογισμούς. το αντίστοιχο προς την υπερβολική και ανώφελη αυτή επιβάρυνση μέρος του δημόσιου χρέους είναι επονίδιστο χρέος το οποίο δεν μπορούν να καλούνται να το πληρώσουν οι πολίτες μέσω περικοπής κοινωνικών δαπανών η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για όλα αυτά και να αποδεχθεί το λογιστικό έλεγχο του χρέους και τη διαγραφή του του μέρους του μέσα από τη σύγκληση μιας πανευρωπαϊκής διάσκεψης για το χρέος. Ο κύριος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τις τελευταίες μέρες μιλήσαμε πάρα πολύ για το ζήτημα της τρομοκρατίας, για το ζήτημα των απειλών κατά της δημοκρατίας. Υπάρχει όμως και μια άλλη απειλή. Μια ασθένεια θα έλεγα, το γεγονός ότι δεν, δεν εμπιστευόμαστε πλέον οι μεν τους δε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να εμφυσίσουμε νέα εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους πολίτες στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και για αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων, να ασχοληθούμε με τα πιο σοβαρά ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει μια στρατηγική κατά της διαφθοράς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ακριβώς ποιο κράτος μέρος λειτουργεί σωστά και ποιο όχι οι πολίτες θα πρέπει να ακουστούν περισσότερο μέσω των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να κάνουν τι απαραίτητε τροποποιήσει στην νομοθεσία τους. Ο κύριος έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Τζοβάνι Φαλκόνε, δικαστής και ήρωας της Σικελίας, έλεγε ότι αν ακολουθήσετε την πορεία των χρημάτων θα βρείτε και τις μαφιόζικες οργανώσεις. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει σημείο κίνησης. Η μαφία αποτελεί παγκοσμιοποιημένο πλέον φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες αναπτύσσονται πιο γρήγορα και από τις ίδιες αγορές. Είμαι από τη Σικελία και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν ήμουν μικρό ότι θεωρούσαμε ότι η μαφία είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει μόνο με το Παλέρμο ή το Κορλεόνε. Ενώ ουσιαστικά ήδη βρισκόταν στη Βόρεια Ευρώπη και στο Μιλάνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η μαφία βρίσκεται στο Παρίσι, στο Λονδίνο, το Βερολίνο πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά, με απόλυτο συντονισμό και απευθύνομαι προς τον Επίτροπο κύριο Βραμόπουλο προκειμένου να λάβει μια σχετική δράση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φεγόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ερμηνεύω το οργανωμένο έγκλημα με τον τρόπο με τον οποίο το κάνει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τραγικές εξελίξεις στη Γαλλία δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από την καταπολέμηση της ε, διεθνούς εγκληματικότητας. Ε, οι τρεις δολοφόνοι αλλά και οι προηγούμενοι εξ αυτών στην υπόθεση Μερά ουσιαστικά ε, πριν ε, γίνουν υπέρμαχοι του ε, Ισλαμισμού ήταν γνωστοί ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι πράγματα που βλέπουμε και στο εξωτερικό με τον Μπόκο Χαράμε, με το Ισλαμικό κράτος και το καθεξής. Δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί και βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα διαδίδονται. Ενδεχομένως η συνθήκη του Σέγγεν είναι ελληματική. Σε κάθε περίπτωση ε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριος Μαλίνοφ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε τι στοιχίζει η διαφορά και το οργανωμένο έγκλημα στις ευρωπαϊκές οικονομίες και τους ευρωπαίους πολίτες. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό, κάτι που δεν μετριέται και αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Η αντίληψη ε, της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος που ε, ε, αναπτύσσονται καταστρέφει την εμπιστοσύνη στους πολίτες. Η δημοκρατία όμως εξαρτάται ε, σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι και μάχη υπέρ της ποιότητας της δημοκρατίας και του μέλλοντος της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη και να την κερδίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, συνενώντας τις προσπάθειες όλων των ε, θεσμικών οργάνων και δεν εννοώ μόνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό, ε, τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, εννοώ και μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών και μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οικονομικών Πληροφοριών που θα αποκαταστήσουν όχι μόνο την εμπιστοσύνη αλλά θα δημιουργήσουν και ένα αίσθημα ασφάλειας. Ως Βούλγαρος Ευρωβουλευτής πρέπει να πω ότι η Βουλγαρία και να ομολογήσω ότι η Βουλγαρία έχει τον υψηλό, από τους υψηλότερους δείκτες διαφθοράς και χαμηλή ε, εμπιστοσύνη στο δικαστικό σώμα. Γι' αυτό εύχομαι ό,τι καλύτερο στις μεταρρυθμίσεις στη χώρα μου. Λόπες Αλγιλάρ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε κύριε Αβραμόπουλε, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνειδητοποιήσει πόσο απαραίτητο είναι να ε, καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξεπλήμα χρήματος. Δεν χρειάζεται να τα συνειδητοποιήσουμε αυτά, τα έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ και χρόνια. Τώρα πρέπει να δράσουμε και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για να υιοθετηθεί κοινό στάνταρ ορισμός του τι εστί οργανωμένο έγκλημα τι εστί νομιμοποίηση παράνομων προσόδων, τι εστί καταπολέμηση παραποιημένων ε, προϊόντων, τι σημαίνει ε, κυβέρνο έγκλημα. Η προστασία των οικονομικών ε, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ξεπεράσει το εμβριακό στάδιο και να γίνει μια πραγματική ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή για να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος, να υπάρξει πλήρη διαφάνεια, για να ε, έχουμε δημόσιο αρχείο όλων αυτών των τραστ και των ε, υπηρεσιών που διαθέτουν στοιχεία και πληροφορίες για τους δικαιούχους και για τους διαμεσολαβητές. Έτσι οι εθνικές αρχές θα συνεργαστούν καλύτερα και θα καταπολεμήσουν καλύτερα το οικονομικό έγκλημα που δεν γνωρίζει σύνορα αλλά και τη διαφθορά. Και θέλω να πω και το εξής φθορά, το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματο απειλεί όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα τη Ένωση, αλλά και την δημοκρατία, τι δημοκρατικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλούν αυτά τα πράγματα την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κόσμου στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι και δημοκρατικό. Θα πρέπει η απάτη να διώκεται, θα πρέπει η παραοικονομία να καταπνίγεται γιατί έτσι θα έχουμε πόρους όχι μόνο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας επιτέλους της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Δεν βλέπω τον κύριο Ρόπε. Η κυρία Κλούν, λοιπόν, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω για το οργανωμένο έγκλημα. Ένα πράγμα μπορούμε άμεσα να κάνουμε όλοι είναι να επιταχύνουμε την οδηγία PNR. Αναφέρθηκε και συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι το οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται πίσω από τις δολοφονίες της περασμένης εβδομάδας στο Παρίσι. Ε, πρέπει λοιπόν να δράσουμε από κοινού τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συμμεριζόμεθα τις πληροφορίες, να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε επίπεδο κρατικό και να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την οδηγία που είναι ζωτική για τον εξοπλισμό των υπηρεσιών ασφαλείας μας για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Το οργανωμένο έγκλημα πλήττει την κοινωνία είτε με τα ναρκωτικά ή την ε, εμπορία όπλων, την εμπορία ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σοβαρές οι μορφές αυτές του εγκλήματος και πρέπει λοιπόν και με μεγάλη σοβαρότητα να τις αντιμετωπίσουμε εμείς ώστε να διατηρήσουμε τις αξίες μας ε, που μεταξύ αυτών την προστασία των ανθρώπων. Επίσης η πορνογραφία, το κυβερνοέγκλημα είναι μεγάλες προκλήσεις, η σεξουαλική ε, κακοποίηση παιδιών online ε, είναι ένα φρικτό έγκλημα και πρέπει να φροντίσουμε οι διαδικτυακές εταιρείες να αναλάβουν την ευθύνη τους και να παίξουν το ρόλο τους ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε από κοινού το κυβερνοέγκλημα. Ευχαριστώ. κυρία Γκόμες έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ο Πορτογάλος Αγγελέας τον Δεκέμβριο του 2014 μετά από 9 χρόνια ερευνών κατέληξε σε αποφάσεις όσον αφορά αγορά συγκεκριμένων υποβρυχίων. Ο Πορτογάλος λοιπόν η συγγελέα είπε ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη συνεργασία από τους Γερμανούς συναδελφούς οι οποίοι ουδέποτε στείλαν τελικά στην Πορτογαλία τα αποδεκτικά εκείνα στοιχεία τα οποία θα είχαν βοηθήσει τις πορτογαλικές αρχές. Ανάλογα πράγματα έχουν συμβεί και στην Ελλάδα με την αγορά υποβρυχίων, ενώ μπορούμε να πούμε ότι είχαν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις στη Γερμανία. Για ποιο λόγο η Γερμανία αυτή τη στιγμή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και νομίζω κύριε Αβραμόπουλο ότι πρέπει να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά οι εγκληματίες όσοι ξεπλέουν μαύρο χρήμα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούν για να νομοποιήσουν τις ε, προσόδους τους. Τι ακριβώς γίνεται λοιπόν προκειμένου να να πατάξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Διακόπτη Πρόεδρος, ο κύριος Μαραγκάλ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα ακούσαμε πληροφορίες για μια αποτυχία συλλογική για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Θα πρέπει όμως να διαλέξουμε να καταπολεμήσουμε τις αιτίε ή να συνεχίσουμε να ε, θεραπεύουμε τα δυσμενή αποτελέσματα. Δεν πρέπει να περιπλέξουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχει όμως κενό νομοθετικό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να έρθει η Ευρώπη να το καλύψει και δεν έχουμε προβληματιστεί ε, επ' αυτού. Το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά, ας το πούμε ξεκάθαρα, είναι ε, προϊόντα της απορρίθμισης του παγκοσμίου ε, οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάτι το οποίο συνέβη πριν από 30 χρόνια. Δημιουργήθηκαν, γεννήθηκαν πριν από 30 χρόνια και ανδρώθηκαν και μετατράπηκαν σε τέρατα τα οποία ε, υπονομεύουν το σύστημά μας, μάλιστα απολαμβάνοντας πλήρη ασυλία. Και θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Η πρόεδρος διακόπτει. Δεν έχετε άλλο χρόνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Προχωράμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Πόλς από ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες ε, συνθήκες οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές κατά την άποψή μου, κάποιες ε, ιδιαιτερότητες. Σίγουρα το οργανωμένο έγκλημα απειλεί την ασφάλειά μας και η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση ε, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Είπατε ότι υπάρχουν 3.000 ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Αυτό το νούμερο είναι πολύ σημαντικό και μας δυσκολεύει ιδιαίτερος. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω και την ε, κακή αξιοποίηση αν θέλετε, των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον. Ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών πολύ συχνά ξεφεύγουν από τα εσκαμένα και πλήττουν ε, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δει αυτό το θέμα. Ο κύριος Νεγκρέσκου για ένα λεπτό. Σίγουρα το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά δεν γνωρίζουν σύνορα και δεν γνωρίζουν και πολιτικό χρώμα αν θέλετε, αλλά βασίζονται στα αδύναμα σημεία της κοινωνίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να υποστηριχθεί ο δικαστικός κλάδος στην Ευρώπη, να στηρίξουμε όλους αυτούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ε, στο ε, σύστημα των διοκτικών και δικαστικών αρχών. Τυρίζουμε ισχυρές ε, ε, δικαστικές αρχές στην Ευρώπη έτσι ώστε να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Θέλουμε η πολιτική να είναι πιο αξιόπιστη, οι πολίτες να συμμετάσχουν περισσότερο, αλλά για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε ελπίδα, να αρχίσουν να πιστεύουν τη δικαιοσύνη. Ε, να, ε, να καταστήσουμε σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη και ότι κανείς διεφθαρμένος δεν έχει θέση στην κοινωνία. Ευχαριστώ. επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ξέρετε, η διακήρυξη ανθρωπίνων όντων είναι ένα από τα πιο αποτρόπαια ε, εγκλήματα. φέρονται τους ανθρώπους έτσι όπως θα φέρονταν σε ένα σακί πατάτες είναι δύσκολο να έχουμε ακριβή στοιχεία για τη ε, λαθρεμπόριο ανθρώπων. Τα θύματα ε, προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης για αδικήματα τα οποία τα εξανάγκασαν να διαπράξουν αντί να θεωρούνται θύματα. Έχουμε την οδηγία κατά του τράφικιν βεβαίως και έχουμε ε, ένα συντονιστή ο οποίο είναι πραγματικά αφιερωμένο ε, σε αυτό το σκοπό, αλλά λίγα γίνονται στην πράξη. Οι κοινέ ερευνητικέ ομάδες, η συνεργασία η διασυνοριακή, η αστυνομική, η βοήθεια της Europol είναι όλα απαραίτητα αλλά όχι αρκετά. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπου έτσι ώστε να βλέπουν τα σημάδια και να τα αναφέρουν για να καταπολεμήσουμε αυτό το έγκλημα το οποίο είναι διασυνοριακό και εξαιρετικά περίπλοκο ήδη από τη φύση του. Η κυρία Αριέλ Γκουσμάν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι περίεργο το ότι Όσοι γνωρίζουν περισσότερα για τη διαφθορά που είναι οι βουλευτές του ΕΛΚ της Ισπανίας, του Λαϊκού Κόμματος, είναι κρίμα λοιπόν που δεν πήραν το λόγο γιατί θα είχαν πολλά να μας διδάξουν. Έχουμε τουλάχιστον χίλιες υποθέσεις ε, ανοιχτές για θέματα διαφοράς, 500 κατηγορούμενους και μία, 20 περίπου στη φυλακή. Και όλα αυτά τα σκάνδαλα έχουν να κάνουν με το Λαϊκό Κόμμα κυρίως, αλλά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα βεβαίως είναι πολύ παρόν. Ε, και ε, η Ευρώπη κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Ενώ το, ε, το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία το μόνο που κάνουν είναι να ε, απογυμνώνουν τον Ισπανικό λαό από την περιουσία του. Μη μας λέτε τώρα τα παραμύθια ότι θέλετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά. Το μόνο που κάνετε είναι να την επιβραβεύετε. Βάλατε για επίτροπο τον κύριο Κανιέτε από το Λαϊκό Κόμμα και βάλετε, ε, βάλατε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον ακατανόμαστο κύριο Γιούνκερ. Ευχαριστώ pour conclure le Κύριος Βαλή και ολοκληρώνουμε τη δικασία catch Ένα λεπτό έχετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω καταρχάς τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, καθώς επίσης και την αρμόδια Υπουργό της Λετωνικής Προεδρίας. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που συμφωνούν. Πρέπει να καλύψουμε τα νομοθετικά κενά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ιταλία. Ξέρετε ότι συνέβησαν διάφορα πράγματα με την ε, σιδηροδρομική γραμμή υψηλή ταχύτητα, τη λεγόμενη ΤΑΒ, όπου είχαμε ένα υψηλό επίπεδο διαφθορά όσον αφορά τι σχετικέ δημόσιε συμβάσει. Ο κύριο Καντών, υπεύθυνο για την καταπολέμηση τη διαφθορά, είπε ότι τα έργα αυτά που συνδέονται με το δίκτυο αυτό υπόκεινται τελικά σε γαλλικό δίκαιο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να διωχθούν από τι Ιταλικέ αρχέ οι παράνομε αυτέ πράξει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί μια προώθηση πλέον από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου οι υπεύθυνοι, αυτοί που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις, να μην εκπροσωπούν το οργανωμένο έγκλημα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει και πάλι το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε τελευταία ανάλυση όλοι συμφωνούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα υπονομεύει όχι μόνο τις οικονομίες αλλά και την κοινωνική συνοχή αλλά και την ασφάλειά μας. Αναμφίβολα είναι μια αυξανόμενη απειλή και αυτό μας θέτει ενώπιον των ευθυνών μας. Όμως η Ευρώπη δεν μένει αδρανής. Έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές, έχει συστήσει ε, θεσμούς όπως η Europol, η Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά. Ε, έχει διοριστεί ο συντονιστής για το τράφικινγκ και βέβαια υπάρχει και το κέντρο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κύβερνο Εγκλήματος στους κόλπους της Europol. Και υπάρχει και η ε, νομοθεσία για το κυβερνοέγκλημα που πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Ε, ανέφερα στην αρχή την μεγάλη συνεργασία που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ε, εμείς ενθαρρύνουμε την συνεργασία επίσης μεταξύ των κρατών μελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οργανωμένο έγκλημα ορίζεται από την ε, απόφαση πλαίσιο του 2008 ε, πρόκειται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το μέσον αυτό ποινικοποιεί επίσης αδικήματα που αφορούν στην συμμετοχή σε μία εγκληματική οργάνωση. Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως η μαφία που αναφέρθηκε πολλές φορές κατά τη συζήτηση καλύπτονται από γενικές διατάξεις που προβλέπονται για όλες τις κατηγορίες οργανωμένου εγκλήματος στην, συμφωνία, στην απόφαση πλαίσιο. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει φέτος μια έκθεση για την ε, υλοποίηση της απόφασης πλαίσιο, όπως είπα ήδη. Για να ολοκληρώσω, αυτό που μας ενώνει όλους εδώ και μέσα στην Ευρώπη είναι η αποφασιστικότητά μας να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα ε, σε όλες τις φάσεις του και να δημιουργήσουμε μια ασφαλέστερη Ευρώπη και ένα περιβάλλον πιο αξιόπιστο για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε πίτροπε. Η κυρία Καλίνκα Λουτσέντκιβα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς να σε ευχαριστήσω για τη διεξαγωγή της σημαντικότητας αυτής συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα καταπολέμησης του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς. Επίσης, να σε ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση αυτή, θα ήθελα να απαντήσω κάποια από τα ερωτήματα τα οποία έθεσαν ορισμένοι βουλευτές, η κυρία Βίξτρομ για παράδειγμα, και να σας πω ότι το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά αποτελούν μια συντονισμένη σφαιρική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκός κύκλος πολιτικής ε, περιέχει πλέον την απαραίτητη μεθοδολογία για να καταπολεμήσουμε τα έγκλημα με τρόπο πιο συντονισμένο χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η νέα στρατηγική εσωτερικής ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει ένα ακόμα θετικό βήμα για την ανάπτυξη, τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προασπίζει τι ελευθερίες και δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να ενισχύσουμε το πλαίσιο αυτό δίνοντα όλο και πιο σφαιρικέ απαντήσει, στις προκλήσει εκείνε που τίθενται από τις οργανώσει οργανωμένου εγκλήματο και από τους παράγοντες της διαφθοράς. Το Συμβούλιο θα συνεργαστεί επικοδοματικά για την έγκριση και την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, αγαπητά αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση. Εξ του FDD Έχουμε ένα αίτημα. Ο κύριος Μάρκος Ζουλού θα αποτελεί μέλος της Επιτροπής ΙΜΚΟ στη θέση της κυρίας Νταϊάν Τζέιμς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις. Αν όχι εγκρίνεται